Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, ήθιστε στην ανάληψη των καθηκόντων του, το πρόεδρο του Κοινοβουλίου να ε, εκφωνεί μία ομιλία ενώπιον τη Συνόδου. Όμω, όταν ανέλαβα τα καθήκοντα τον Ιανουάριο, θεώρησα ότι ήταν σκόπιμο να περιμένω κάπω πριν να μοιραστώ μαζί σα το δικό μου άποψη για τα πράγματα. Έτσι μπόρεσα να μετρήσω καλύτερα το βάρος των ευθυνών που φέρω ως Πρόεδρος, αλλά και το βάρος της ευθύνης που φέρουμε όλοι ως ένας θεσμός και ως ε, βουλευτές. Μένουν λιγότερο από δύο έτη πριν τις εκλογές και έχουμε ενώπιόν μας ε, μεγάλες προκλήσεις. Ε, τρομοκρατία, μετανάστευση, παράνομη μετανάστευση, απασχόληση, κλιματικές αλλαγές, Brexit. Οι συμπολίτε μας μας ζητούν να απαντήσουμε στις προσδοκίες τους. Ας απευθύνονται σε εμά προσδοκούν από εμά, γιατί σε ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε οι άμεσοι του συνομιλητέ. Τον Μάρτιο είχα τη τιμή να υπογράψω στο όνομα του Κοινοβουλίου τη δήλωση της Ρώμης, ε, τη δέσμευση να επαληθεύουμε διαρκώς ότι οι στόχοι που έχουν θέσει οι κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν θα μείνουν δηλώσεις προθέσεων, αλλά θα μεταφραστούν σε πραγματικές απαντήσεις ε, για του συμπολίτε μας. Υιοθετήσαμε σημαντικές ε, ρυθμίσεις όπως το ΕΦΣΙ, το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης, ε, το Δέσμι για την Προστασία των Δεδομένων ή ακόμα την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Από τις αρχές του έτους έχουμε κάνει πολλά, σταθεροποιήσαμε τις χρηματοπιστωτικές αγορές, έχουμε ε, φτιάξει την, ε, το Ταμείο ε, Κοινωνικής ε, αρρωγής και σε λίγα λεπτά θα ψηφίσουμε και για μέτρα τα οποία στόχο θα έχουν την ασφάλιση, ε, στην ασφάλεια ανεφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Πολλά ακόμα όμως πρέπει να γίνουν. Θέλουμε αποτελέσματα στα πλαίσια της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Πρέπει να εξυγχρονίσουμε την εμπορική μας πολιτική ώστε να προστατεύσουμε τις στρατηγικές μας βιομηχανίες. Οφείλουμε να, ε, να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να βρούμε μια συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των εκπομπών ε, και να εξασφαλίσουμε την μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια. Η νέα Επιτροπή για τον Τρομοκρατία ασχολείται για το, με το πώς θα βελτιώσει τον αγώνα κατά αυτής ε, της πληγής, να ενισχύσει την άμυνα και να ενισχύσει επίσης την επιμηχανική πολιτική. Το πιο περίπλοκο έργο που μας ε, περιμένει είναι ε, η δέσμοι για το άσυλο. Γνωρίζουμε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στο Συμβούλιο. Ωστόσο, αυτό δεν μας απαλλάσσει από το δικό μας καθήκον να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα για να ολοκληρωθεί η εξέταση αυτού, του, αυτής της δέσμης μέτρων πριν από το πέρας της θητείας μας. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο της Επιτροπής, μας, Επιτροπής όταν θα συζητήσουμε την κατάσταση της Ένωσης. Είμαστε μια, ένας μηχανισμός νομοθετικός εξαιρετικά περίπλοκος, ωστόσο πιστεύω πως λειτουργεί αρκετά καλά και χαίρομαι ε, γιατί γι' αυτό βασιζόμαστε σε μια ικανή, επαγγελματική και αφοσιωμένη διοίκηση. Θα προσπαθήσω να διατηρήσω την αρμονία και την χρηστή συνεργασία ανάμεσα στα διάφορα όργανα του Συγκοινοβουλίου, γιατί από αυτά εξαρτάται η αποτελεσματικότητα και η δυνατότητα δράσης μας. Η απόδοσή μας εξαρτάται επίσης και από τις συνθήκες εργασίας. Γι' αυτό και αποδίδω σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά θα ήθελα ε, να πω ότι αγαπητοί συνάδελφοι δεν υιοθετούμε μια νομοθεσία απλά και μόνο για να μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι κάτι κάναμε στον τάδε δυνατομέα. Έχουμε την υποχρέωση να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις και να προβούμε στις σωστές επιλογές γιατί η νομοθεσία που υιοθετούμε έχει επιπτώσεις στη ζωή 500 εκατομμυρίων πολιτών για τις επόμενες δεκαετίες οι νομοθεσίες θα πρέπει να συζητώνται εις βάθος ε, σε όλες τις πτυχές θα πρέπει να, να ακούμε προσεκτικά τους συμπολίτε μας αλλά και τη συνείδησή μας. Βεβαίως ε, ε, πρέπει να αποφεύγουμε τις μακροχρόνιες καθυστερήσεις και τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και θα μερυμνήσω ώστε αυτοί οι νεκροί χρόνοι να μειωθούν το ελάχιστο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμβάλλει στην υιοθεσία νομοθετημάτων ποιότητα που θα λύνουν τα προβλήματα των πολιτών και να μην δημιουργούν νέα. Όμω ταυτόχρονα οι πολίτε περιμένουν να υπερασπιστούμε στην Ευρώπη και στον κόσμο τι αρχέ μα και τι αξίε μα, την ελευθερία, την αλληλεγγύη, την επικουρικότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την ισότητα ανδρών γυναικών, την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Είμαι πεπισμένο ότι οι πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται εδώ από την ίδια ε, ε, επιθυμία εμπνέονται να βελτιωθεί η κατάσταση διαβίωση των συμπολιτών μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, επίσης ε, έχουμε να κάνουμε τα δύο, είμαστε το ένα από τα δύο σκέλη τη δημοσιονομική αρχή. Πρέπει να αναλάβουμε αυτή μα την ευθύνη όπω ανέκαθεν κάναμε με ένα όραμα αυτή τη στιγμή ξεκινάνε συζητήσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Είμαι πεπισμένο ότι ο νέο προπολογισμό πρέπει να είναι πολιτικό προπολογισμό που να βγαίνει από τι διανεμητικέ λογικέ και να βασίζεται σε σαφεί στόχου. Πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνουν οι πολιτικέ επιλογέ. Και μόνο κατόπιν μπορούμε να αποφασίσουμε του δημοσιονομικού πόρου για να του επιτύχουμε. Όχι το αντίστροφο. Το Κοινοβούλιο έχει, πρέπει να εκφραστεί επανειλημμένα στην ανάγκη για την ανάγκη να υπάρξουν νέοι ήδη πόροι. Είμαι πεπισμένο ότι υπάρχει όντω τέτοια ανάγκη και καλό να συνεχιστεί η συζήτηση στα πλαίσια του σώματός μας και με τα άλλα θεσμικά όργανα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κοιτάξτε γύρω σας το σώμα μας. Σε αυτό το ημικύκλιο έχουμε συναδέλφους από όλες τις περιοχές της Ευρώπης, από τις γωνιές τις πιο απομακρυσμένες της Υπήρου μας, και ακόμη και από τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Εδώ εκπροσωπούνται όλοι οι λαοί τη Ένωση. Το κοινοβούλιο μας είναι, είναι η καρδιά της Ευρώπης. Το κοινοβούλιο είναι ο μόνος χώρος στην Ήπειρό μας όπου οι άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι μπορούν να συζητήσουν ανοιχτά θέματα που αφορούν ολόκληρη την Ήπειρο. Ο μόνος χώρος όπου μπορούν να αντιπαρατεθούν, να γνωριστούν και να συνεργαστούν για να επιλύσουν τα κοινά προβλήματα. Στο σώμα μας έχουν εκφραστεί αρχηγοί κρατών, των κρατών μελών και του κόσμου όλου και διακεκριμένες προσωπικότητες ε, μεγάλες προσωπικότητες της εποχής μας. Αυτό αποδίδει στο σώμα μας μια διάσταση που ξεπερνά κατά πολύ το ρόλο που, τις αποδίδουν, που του αποδίδουν οι συνθήκες. Αυτή η διάσταση πρέπει να ενισχυθεί. Οπότε θέλω να υπενθυμίσω, ε, δράτω με τις ευκαιρίες για να υπενθυμίσω σε όλους τους αρχηγούς κρατών, των κρατών μελών της Ένωσης, ότι έχουν μόνιμη πρόσκληση για να εκφραστούν στην Ολομέλειά μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε μια ανεκτήμητη πληθώρα ιδεών και πολιτικών ευαισθησιών και ε, απόψεων. Θέλουμε φυσικά να μπορούμε να συζητάμε στο κοινοβούλιο, αλλά μόνο με βάση ιδέε και αμοιβαίου σεβασμού. Είμαστε ένα ζωντανό κοινοβούλιο και θα κάνω ό,τι μπορώ, ούτω ώστε όλε οι ενέργειε και οι ιδέε που εκπροσωπούνται σε αυτή την αίθουσα να μπορέσουν να εκφραστούν και να συμβάλλουν στη συζήτηση και στην σκέψη. Όπω λέω πάντα, θέλω να είμαι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου. Δεν θέλω να είμαι ένα πρωθυπουργό το Κοινοβούλιο πρέπει να ηγηθεί εκ νέου για τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και να δώσει την πολιτική όθηση που χρειάζεται μόνιμα η Ένωση. Πρέπει να αλλάξουμε την Ευρώπη εκεί που χρειάζεται. Αλλά πρέπει να επιτευχθεί πρόοδο. Ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που τον ευχαριστώ, μα υπέβαλε ένα σύνολο ιδεών για το κοινό μα μέλλον. Ξέρω ότι όλε οι πολιτικέ οικογένειε συζητούν αυτό το θέμα. Ήρθε η ώρα να ανταλλάξουμε τα απορίσματά μα. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μια μεγάλη ανοιχτή συζήτηση στην Ολομέλεια. Επίση θα πρέπει να ανταλλάξουμε απόψει με του άλλου βασικού ευρωπαϊκού φορεί και προσωπικότητε που πρέπει να προσκαλέσουμε. Αυτή θα είναι μια ευκαιρία ούτω ώστε να είμαστε στο επίκεντρο τη συζήτηση και να παίξουμε το ρόλο φόρουμ πολιτικών συζητήσεων που είναι ακριβώ ο ρόλο μα, αγαπητοί συνάδελφοι. Κατά την ε, εναρκτήρια ομιλία τη, ε, η διακεκριμένη Προκάτοχό μου, η κυρία Σιμών Βέιλ, υπενθύμησε ότι ο δημοκρατικό έλεγχο είναι η πρώτη λειτουργία κάθε εκλεγμένη συνέλευση. Πρέπει λοιπόν να είμαστε απαιτητικοί στην ε, άσκηση αυτού του ελέγχου έναντι τη εκτελεστική εξουσία. Η πρακτική των επικεφαλών των επικεφαλής ψηφοδελτίων, των Spitzenkandidaten, ενισχύει την εμπιστοσύνη μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να εδραιωθεί αυτή η εξέλιξη. Για να λειτουργήσει η Ένωση, η Επιτροπή πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τη στήριξη του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, αυτή η εμπιστοσύνη δεν είναι αυτόματη. Πρέπει να κερδίζεται κάθε μέρα. Επίσης είμαι υπέρ της καλής συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, του αμοιβαίου σεβασμού, της έντιμης συνεργασίας. Η ένωσή μας είναι η δύναμή μας, να μην το ξεχνάμε ποτέ. Η ιστορία μας καταδεικνύει ότι η ενίσχυση της Ένωσης πάντα συνοδεύτηκε με την ενίσχυση του Κοινοβουλίου. Παραμένω πεπισμένος ότι η μάχη για να αποκτήσουμε ένα δίκαιο πρωτοβουλία είναι θεμελιώδης. Προς αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να συνεχιστεί. Η ενίσχυση της ε, κοινοβουλευτικής διάστασης της Ένωσης περνά επίσης μέσω όλο και πιο στενής συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια. Η Ευρώπη είτε θα είναι δημοκρατική είτε θα υπάρξει και επιμένω, το Κοινοβούλιο είναι η ζωντανή καρδιά της δημοκρατίας και δίνει δημοκρατική νομιμοποίηση στην Ένωση. Χωρίς το Κοινοβούλιο, η Ένωση θα ήταν ένα σύστημα συνεδριάσεων με μια ε, ψυχρή γραφειοκρατία. Το Κοινοβούλιο διασφαλίζει την υπεροχή της πολιτικής έναντι της γραφειοκρατίας Και το Κοινοβούλιο είναι επίση το ηχείο των προσδοκιών των συμπολιτών μας. Πρέπει να του ακούσουμε. Πρέπει να έχουμε έναν μόνιμο διάλογο ανοιχτό και διαφανή μαζί του. Είμαστε το πιο ανοιχτό κοινοβούλιο στον κόσμο. Κάτι τη διάρκεια τη θητεία μου θα κάνω ό,τι μπορώ, ούτω ώστε οι πόρτε μα να είναι ανοιχτέ για του συμπολίτε μα. Κάθε βουλευτή καλείται να παίξει θεμελιώδη ρόλο σύνδεση μεταξύ των πολιτών και των θεσμών τη Ένωση. Δεν είναι μόνο εκπρόσωπο ε, των πολιτών έναντι της Ένωσης, αλλά είναι και εκπρόσωπο της Ένωσης έναντι των πολιτών. Είναι πολλή δουλειά αυτή και μας απασχολεί κάθε στιγμή του χρόνου μας και τα Σαββατοκύριακα. Γι' αυτό πρέπει να πούμε δυνατά ότι οι βουλευτές δεν είναι μόνο το δάχτυλο στην μηχανή ψηφοφορίας, είναι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού λαού, πρέπει να το σεβαστή. πρέπει να ακούγεται η φωνή τους. Είναι, έχουν φωνή και πρέπει να ακούγεται. Αυτό είναι το όραμά μου και θα κάνω ό,τι μπορώ ούτω ώστε η αξιοπρεπία των βουλευτών να διατηρηθεί και ο ρόλο του να αξιοποιηθεί. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό που είμαστε. Εγώ και ω πρόεδρο, αλλά και ω συνάδελφό σα, είμαι περήφανο για την εργασία σα εδώ και εκτό αυτού του ημικυκλίου. Σα ευχαριστώ για αυτά που γίνονται στου διαδρόμου, στι επιτροπέ, στι πολιτικέ ομάδε, στα διάφορα όργανα του σώματο και κυρίως ενώπιον των εκλογέων σας. Σα ευχαριστώ για την ε, ενέργεια που δαπανάτε κάθε μέρα στις συζητήσεις, στις διαπραγματεύσει, τις ε, συναντήσεις, τις επαφές με τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών. Η εργασία σας δεν είναι πάντα τόσο ορατή, αλλά τελικά αυτή διασφαλίζει την λειτουργία της δημοκρατίας στα πλαίσια τη Ένωση. Είμαι περήφανο για εσά. Είμαι περήφανο που είμαι πρόεδρο αυτού του Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστώ επίση. Σας ευχαριστώ επίσης για την εμπιστοσύνη που μου χορηγήσατε. Θα κάνω ό,τι μπορέσω για να ανταποκριθώ σε αυτήν. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Χαίρετε αγαπητοί συνάδελφοι και σε αυτό το ευχάριστο φιλικό κλίμα περάσουμε στις ψηφοφορίες. Αλλά κάποιος ζήτησε το λόγο για διαδικαστικό, αν δεν κάνω λάθος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ενημερώσω το, την Ομιγύρη ότι χθε ε, μια νεαρή Ισπανίδα, η Λορένα Νευράλ, δολοφονήθηκε ενώ ασκούσε το έργο της ε, στο Αφγανιστάν, στον Ερυθρό Σταυρό. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλει ένα μήνυμα στήριξη και αλληλεγγύη προ την οικογένεια τη ε, νεαρή Ισπανίδα, τον Ερυθρό Σταυρό και την αναγνώρισή μα προ του άνδρες και τι γυναίκε που αφιερώνουν τι γνώσει του το χρόνο και τη ζωή του μερικέ φορέ ε, στην βοήθεια των συνανθρώπων του Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε και για τις αντιδράσεις. Έχουμε 50 περίπου ψηφοφορίες ενώπιόν μας. Ας φροντίσουμε λοιπόν.